αφορά το Σουδάν και την περίπτωση του δόκτωρος Αμίν Μέκη Μεντάνη. Το λόγο έχει η κυρία Σαρζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητούμε ε, να δοθεί η απαραίτητη προσοχή σε τρεις ε, ακτιβιστές, τον κύριο Φαρούκ Αμπού Ισά, τον κύριο Φαράχ Ιμπραήμ Μοχαμέτα Λαγάρα ε, και τον δόκτωρα Αμίνε Μεκί Μεντανή θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όπως ε, το κάναμε και για την πρόσφατη περίπτωση της Σουδανής που ήταν φυλακισμένη με το παιδί της. Ο κύριος ε, Αμίν μεκή ε, Μεντανή συνελήφθη στο Χαρτούμ την πρωτεύουσα του Σουδάν επιστρέφοντας από εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα είναι αυθαίρετη και η σύλληψη και η κράτηση του δόκτωρος ε, Μεντανή ε, διότι ε, απλώς συνελήφθη διότι μιλούσε υπέρ της ε, αντιπολίτευσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μελετηθεί από κοντά η κατάσταση σε μια χώρα σαν το Σουδάν γιατί διαρκώς τα πράγματα αλλάζουν ε, και ε, διαρκώς η πίεση και η βία αυξάνει από την κυβερνητική πλευρά και τις κυβερνητικές δυνάμεις. Θα πρέπει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητήσουν ε, ε, με την, ε, με την Αφρικανική διάσκεψη έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα. Αλλά τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια να συζητηθούν τα προβλήματα των χωρών βλέπουμε σκανδαλώδεις συλλήψεις όπως αυτές του δόκτωρα Αμίν Μεκί Μεντανή, του Φαρούκα Μπουισά και του Φαράχ Ιμπραχήμου Ταμέδα Λαγάρ. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν δια της βίας στη χώρα. Ησυχία παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Έλερ. Πρόεδρε, αγαπητοί της συνάδελφοι, τον Μάιο φοβηθήκαμε, τρομάξαμε από την ε, θεραντική καταδίκη της Ιμπραΐσικα η οποία θα ε, το, θα ε, έχανε τη ζωή της, αλλά τελικά φροντίσαμε να απελευθερωθεί. Τώρα λοιπόν ε, ο Αμιν Μέκη Μεντάνη χρειάζεται την προσοχή μας. Ε, είναι ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν και στις 6 Δεκεμβρίου συνελήφθη από τις μυστικές υπηρεσίες του Σουδάν ε, διότι υπέγραψε το περίφημο Σούδαν Κόλ όπου πολλοί εκπρόσωποι, πολιτικοί εκπρόσωποι του Σουδάν επισημαίνουν την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές περιοχές του Σουδάν και ε, ζητούν τη διαδικασία της ε, συμφιλίωσης. Εμείς λοιπόν ζητούμε, απαιτούμε την πάραυτη απελευθέρωση ε, του γιατρού, ο οποίος είναι ήδη 76 ετών και χρειάζεται απαραίτητα φάρμακα, κάτι που δεν του το δίνουν οι αρχές του Σουδάν. Αυτό λοιπόν είναι μια απειλή για τη ζωή του και γι' αυτό ζητάμε από τις αρχές του Σουδάν επιτέλους να δρομολογήσουν ειρηνική διαδικασία και να σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα τους. Ο κύριος Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, ε, το ECR καλεί τις αρχές του Σουδάνα ε, να ελευθερώσει τον δόκτωρα Αμίν Μέκη Μεντάνη και όλους τους υπολείπους ακτιβιστές ε, άμεσα. Είναι ένας νόμιμος ακτιβιστής υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ζωή του αυτή τη στιγμή απειλείται. Είναι 76 χρονών, πάσχει από διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση και δεν του δίνουν τα φάρμακά του εμ Επίσης, ο Μαραλ Μπασίερ δεν έχει δυστυχώς λάβει θέση ε, όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να σταματήσουν όλες οι διώξεις αλλά και η η αντιμετώπιση και η τρομοκράτηση όλων των ακτιβιστών ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα που συζητούμε για το Σουδάν και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. Και πολλές φορές επειδή μας ενδιαφέρει η σταθερότητα δεν θα πρέπει να μελούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί η σταθερότητα νοείται μόνο όταν ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκκληση για το Σουδάν, το Sudan Call. Αυτό ακριβώς προβλέπει και οι προσυπογράφοντες ε, μαζί με τον ε, δόκτορα Μεντάνη. Ε, αυτό ακριβώς το θέμα δήλωναν μαζί με άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης. Ζητούμε άμεση απελευθέρωση του δοκτώρος Μεντάνη και την συνέχιση του διαλόγου με τις επικοδομητικές δυνάμεις του Σουδάν. Ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσατε να γίνεται λόγος ε, για αυτήν την έκκληση Σούνταν Κόλ. Ε, είναι έκκληση και συλλογή υπογραφών για να σταματήσει αυτή η τακτική του ενός κόμματος ε, στο Σουδάν αλλά ε, αυτού του είδους ε, η διαδικασία σταμάτησε όταν ε, άρχισαν οι μυστικές υπηρεσίες να συλλαμβάνουν τους υπογράφοντες όπως τον δόκτωρα Αμίν Μεκί Μεντάνη, τον Φαρούκ Αμπού Ισά και άλλους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι φυλακίστηκαν διότι είχαν αντιταχθεί στην κυβέρνηση του Σουδάν. Καθημερινά υπάρχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ανθρώπων και ε, φυλακίζονται όσοι ειρηνικά προσπαθούν να αντιταχθούν. Είναι ένα καλό ψήφισμα και πρέπει να περάσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέιτ. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στο Σουδάν χρήζει προσοχής. Ε, έχουμε συνεχείς αναφορές για βασανιστήρια και διώξεις ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρήση σεξουαλική βία από πλευρά ε, ε, ε, στα στρατιωτών, ακόμη και ομαδικούς βιασμούς νεαρών κοριτσιών θα πρέπει το Σουδάν να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις και τις προδιαγραφές ε, διεθνώς, όπως και την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και όλα τα εργαλεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν ε, κυρωθεί από το Σουδάν. Η πρόσφατη προ... Ε, σύλληψη του, δοκτώ... του Μεντάν είναι άλλο ένα παράδειγμα του τι πάει στραβά στο Σουδάν. Ζητούμε άμεση αποφυλάκηση. Και μάλιστα η εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατέθεσε τεκμήρια για διάπραξη γενοκτονία γενοκτονίας, ε, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου από πλευρά Πρόεδρου Αρμπασίρ, ο οποίος συνεχίζει να κρατά τα ενία τη εξουσία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει αυτό που αποφάσισε και να ζητήσει άμεση ε, διακοπή τη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν και την συνεχιζόμενη δίωξη ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Βεριζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι από αυτούς ε, και μεταξύ αυτών που καταδίκασαν χτε ε, την διαδικασία του Χαρτούμ ε, και για το κέρα της Αφρική. Η κατάσταση από το 2009 διαρκώς χειροτερεύει στο Σουδάν. Αλλά ποτέ δεν είχαμε τέτοια συγκέντρωση της αντιπολίτευσης. Πράγμα που εξηγεί και την βιαιότητα με την οποία αντιδρά η Σουδανική κυβέρνηση. Έχουμε βομβαρδισμούς αμάχων, έχουμε ε, βίαιη ομή καταστολή προς κάθε κατεύθυνση. Ε, η ε, Αμίνε Μεκί Μεντανή, Φαρού Καμπού Ισά και Μοχαμέντα Λαγάρ είναι σύμβολα πλέον. Είναι ασυγχώρητη η στάση και των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν καταφέρει να καταδικάσουν αυτές τις πράξεις. Θα πρέπει αμέσως να ελευθερωθούν οι θα πρέπει να στηρίξουμε ε, τον λαό του Σουδάν έτσι ώστε να μπορέσουν να ζήσουν με ειρήνη και όχι σε κατασταλτικά δικτατορικά καθεστώτα. Γκαμπούς. Ευχαριστώ κύριε Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι μιλώ σε ένα δημόσιο βήμα όπως τώρα. Δεν θα χρησιμοποιήσω το χρόνο μου συνοψίζοντας τα πραγματικά περιστατικά γιατί τα γνωρίζουμε. Ο δοκτώρ Αμίν Μεντάνη φαίνεται ότι είναι επικίνδυνος άνθρωπος. 76 ετών είναι άνθρωπος, έχει ιατρικά προβλήματα, είναι άρρωστος. Αλλά συνελήφθη μαζί με άλλους και άλλες που θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για το λαό του και μάλιστα διαδήλωσαν ειρηνικά, ε, διεκδίκησαν αυτό το μέλλον με δημοκρατικούς τρόπους, με τα δικαιώματα των πολιτών και με βάση αρχές που ενστενιζόμαστε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αναλαμβάνει κανείς δράση ζητώντας την, τον των ένοπλων σειράξεων στο Σουδάν και τη θέσπιση των απαραίτητων θεσμικών, νομικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Είναι κρίσιμη η κατάσταση στο Σουδάν, πολύ εύθραυστος ο πολιτικός διάλογος, γι' αυτό και η συμβολική παρουσία του κυρίου Μεδάνη στο πολιτικό προσκήνιο είναι σημαντικότερο από ποτέ. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση του Σουδάν να εξασφαλίσει ε, ειρηνική άσκηση των δικαιωμάτων, το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης ε, του συνέρχεστε και του συναθρίζεστε και άμεση αποφυλάκηση των υπερμάχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δόκτωρος Μεντάνη και άλλων. Η κυρία Κέγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι άνεμοι του πολέμου στο Σουδάν δεν έχουν κοπάσει. Έχουμε διαρκώς και σε ολόκληρη τη χώρα παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλονται από, τους, ε, ε, από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Οι βομβαρδισμοί στο Ταρφούρ, ε, οι, οι ομαδικές καταγγελίες που έχουμε όσον αφορά τις επιδρομές κατά αμάχων στον Κιανού Νείλο, οι επιθέσεις στο Νότιο Κορντοφάν είναι μερικές από τις περιπτώσεις τις οποίες πρέπει να καταγγείλουμε και που καταγγέλλονται από διαφόρους ε, Σουδανούς ε, φωνές ε, οι οποίες ακούγονται όλο και περισσότερο μεταξύ των οποίων αυτή του Αμίν Μεκί Μεντανή και άλλων. Μέσω του ψηφίσματος αυτού κύριε Πρόεδρε ζητούμε με τεπιτάσεω να ξεκινήσει συνολικός διάλογος για την ειρήνη έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα να γίνει κράτος δικαίου και πραγματική δημοκρατία γιατί διαφορετικά όλη η περιοχή του κέρατος της Αφρικής πολιτικής κινδυνεύει ε, να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα όχι μόνο στην Αφρική αλλά και σε άλλες πλευρές του κόσμου μέσω μαζικών μεταναστευτικών κυμάτων. Κυρία και δεν έχετε άλλο χρόνο. Κύριο Στομασεύσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στο Σουδάν γίνεται όλο και πιο ασταθής. Και μάλιστα το Σουδάν φτάνει σε ένα σημείο καμπής στην ιστορία του. Οι δημόσιες αρχές εφαρμόζουν ε, βάναυσες ε, και κατασταλτικές ενέργειες αστυνομικού κράτους, παράνομες δραστηριότητες κατά των ακτιβιστών είναι δραστηριότητες και ενέργειες που καταπατούν τα διεθνή δικαιώματα και τις διεθνείς τα διεθνώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς προδιαγραφές. Για παράδειγμα η σύλληψη του δόκτωρο Σαμίν Μέκη Μεντάνη σημαντικού υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του λαού του Σουδάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει και ε, να επισημάνουμε την ανάγκη σεβασμού και της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Δεν μπορεί η θρησκευτική πίστη να είναι λόγος για δίωξη. Θα πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό και απερίφραστο μήνυμα. Είμαστε κατά των διακρίσεων. Παρακαλώ, ησυχία. Σας θέρμο παρακαλώ. Ησυχία. Ο κύριος Καστάλντο Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το Σουδάν και όλα είναι οδυνηρά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νταρφούρ. Ε, Μία κρίση η οποία εδώ και χρόνια υπάρχει και η οποία δεν ε, φαίνεται να είναι έτοιμη να σταματήσει. Μπορούμε να μιλήσουμε για εγκλήματα πολέμου ε, στην περιοχή. Αλλά βλέπουμε ότι ο Αλβασίρ βρίσκεται πάντα στη θέση του και ότι δεν γίνεται τίποτα καλύτερο. Και επομένως σπαταλούμε μάταια τους τους πόρους μας. Θα ήθελα εδώ να κάνω μία έκκληση ε, για τον δόκτωρα Αμίν Μεκί Μεντάνη, έναν θαραλέο άντρα, παρότι ηλικιωμένο και άρρωστο. Ε, είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε την πολιτική δήλωση Σουντάν Κολ, εξ ονόματος ε, μιας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν το Σουντάν Κολ, δημοσιογράφοι, απλοί άνθρωποι, πολιτικοί, έχουν, είναι πλέον ε, φυλακισμένοι. Πρέπει να επελευθερωθούν. Απελευθερώστε τους. Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση του Σουδάν αλλά και στην διεθνή κοινότητα. Ε, η χώρα, ε, το Σουδάν είναι μια χώρα η οποία φυλακίζει το μέλλον της. Σας ευχαριστώ κύριε Σοπράτ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στις 6 Δεκεμβρίου ο δόκτωρο Αμή Μεκί Μεντανή ε, δικηγόρος ε, ε, και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φυλακίστηκε, συνελήφθηκε, φυλακίστηκε στο Χαρτούμ. Ε, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ε, ζητάει ε, ελευθερία στο Σουδάν. Και εμείς πρέπει να ζητάμε την απελευθέρωση του δόκτωρο Σαμεντανή αλλά και γενικότερη ελευθερία. Ξέρουμε ότι οι θρησκευτικές ελευθερίες καταπατώνται. Ξέρουμε τι έγινε με την χριστιανή Μυριάμ η οποία κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ε, δεχτούμε ε, και ένα, ε, μια κίνηση από πλευράς της δύση που κουνάει το δάχτυλο μπροστά από μια χώρα. Εμείς δεν μπορούμε να υποδεικνύουμε διαρκώς τον δρόμο σε μια κυβέρνηση γιατί και γι' αυτό το λόγο θα απόσχουμε βεβαίως καταδικάζουμε τα εγκλήματα αλλά δεν μπορούμε να συμβάλλουμε σε, αυτά, σε τη διδασκαλία προς χώρες. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Γκέριγκερ, κύριε Πρόεδρε, για μία ακόμη φορά συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα δίωξεων εκ μέρους του Σουδάν ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Στις 6 Δεκεμβρίου συνελήφθη χρονος δόκτωρ Ατμίν Μέκη Μεντάνη, γνωστός ακτιβιστής και υπέρμαχο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ήταν απάντηση στην υπογραφή που έβαλε στην έκκληση για το Σουδάν και την αποκατάσταση κράτους για του πολίτε και τη δημοκρατία μαζί με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως ε, το Σουδανικό Επαναστατικό Μέτωπο που ζητούν ε, κατάπαυση του πυρός και των ένοπλων σειράξεων και ε, θέσπιση των κατάλληλων νομοθετικών, οικονομικών και άλλων μεταρρυθμίσεων. Καταδικάζουμε δρυμύτατα την κράτηση, την παράνομη κράτηση του Μεντάνη που είναι άρρωστος και μάλιστα δεν, δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και επίσης ε, θα πρέπει το Σουδάν να τηρήσει τα, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να εξασφαλίσει την ελευθερία έκφρασης, ε, την ελευθερία του συνέρχεστε και την ελευθερία θρησκευτικής πίστης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως ακούσατε, ε, ο Δόκτωρ Μεντάνη στις αρχές ε, Δεκεμβρίου συνελήφθη από τις αρχές του Σουδάν και εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι ακόμα γνωστό το αίτιο, ίσως ε, και προφανώς διότι υπέγραψε την έκκληση για το Σουδάν, μια πρωτοβουλία η οποία επιθυμεί να φέρει τη δημοκρατία στο Σουδάν. Κατά την άποψή μου τραγικό το γεγονός ότι σλαμβάνεται ένας 76χρονος γιατί τάσεται υπέρ της δημοκρατίας. Στις 14 Δεκεμβρίου αυτού του έτους στην Τουρκία συνελήφθησαν 31 άτομα, 31 άτομα εκ των οποίων πολλοί δημοσιογράφοι και αυτό κατά την άποψή μου ε, πρέπει να το προσέξουμε. Να προσέξουμε το τι κάνει η Τουρκία κυρίως αν έχουμε κατά νου ότι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος επιβαρύνεται κάθε χρόνο με ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Από το 2007 μιλάμε δηλαδή για συνολικά 4,9 δις ευρώ χωρίς υπεραξία των αντίον από ό,τι φαίνεται η Τουρκία εξακολουθεί να, εξακολουθεί να ακολουθεί λάθος δρόμο. Ευχαριστώ. Κανονικά έχουμε catch the αλλά δυστυχώς ε, δεν μπορούμε ε, λόγω έλλειψης χρόνου να περάσουμε στο catch the πριν όμω δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, θα ήθελα να καλωσορίσω μία αντιπροσωπεία της Ελβετικής Βουλή, με επικεφαλή στην Κάτι Ρίκλη και με παρουσία αντιπροέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων του Εθνικού Συμβουλίου, τον κύριο Λάνου Αβεσέλη, ε, της Επιτροπής ε, ε, Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Χριστιαν Λεμπράντ.